πληροφορία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βάσει του άρθρου 231 παράγραφος 4 δεν έχει ζητηθεί ε, ψηφοφορία για το διορθωτικό που αναγγέλθηκε χθε στις 5 το απόγευμα, οπότε το διορθωτικό